Brasilianers. Kolleginnen und Kollegen, darf die Nachmittagssitzung eröffnen. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή μα ε, συνεδρίαση για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση το πρωί. Συνεχίζουμε με το σημείο 10 πάντως της διάταξης προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Ε, κυρία Σεις, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά, κατά αποχές δεκτή. τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Πέρασε. Παρακαλώ επαναλάβετε γιατί είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα το μηχάνημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Περισσεύει ένας από την ομάδα των Άλντι και άλλος ένας από την ομάδα των Πρασίνων. Βέβαια δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει έχει εγκριθεί. Τροπολογία 8. Υπέρ. Με ναι, ανάπτυξη χειρών. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 και 15 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 17 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 17. Πάλι περισσεύουν ορισμένοι βουλευτές. Ένας από το ΕΛΚΑ, ένας από τους φιλελεύθερους, ένας από τους... Πάρα πολύ περισσεύουν. Και ένας πράσινος ακόμα περισσεύει. Κάθε μπορεί να το πει αυτό. Τι γίνεται, γιατί έχουμε τόσους πολλούς. Ο Άλτε, οι Άλτε έχουν ένα παραπάνω ή δεν ψηφίζεται. Είμαστε έξι στην Άλντε και κανονικά πρέπει να είμαστε οκτώ. Δεν μπορούμε να είμαστε πολλοί άμα είμαστε, μάλλον λιγότεροι από ό,τι πρέπει είμαστε. Είναι σχετικό αυτό που λέτε, λέει ο πρόεδρος. Jetzt soll's klappen. Εντάξει, ναι. Τώρα είναι εντάξει, λέει η γραμματεία. Ψηφίζουμε λοιπόν και πάλι. Τροπολογία 17. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29-28 εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για 18 18 πέρας εγκρίνεται 31-22 τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρόπολογια 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές 45 υπέρ Πάλι. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος καλά. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. εγκρίνεται 32, 28. Δέκτη λοιπόν. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. 51 με 10 υπέρ με 10 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. Συγχωρητήρια κυρία Ασής. Περνάμε. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τάνοκ. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι κύριε Τάνοκ. Δεν έχει παρατήρηση. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κάτι έχω λάθος εδώ στον κατάλογό μου. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Να ελέγξουμε την 55. Ίσως βιάστηκα να δώσω το αποτέλεσμα. Πέραση της ψηφοφορία. 26 υπέρ 40 κατά απορρίπτεται. Λοιπόν, 56 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, να ελέγξουμε την 84. Πέραση ψηφοφορία. 30 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε την 102. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 35 κατά, απορρίπτεται. 102, όχι την 102 ψηφίσαμε. 107 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Υπέρ πάλι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 Ψηφίσαμε την 115 πριν, τώρα έχουμε περάσει την 116. 116 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 119 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 36 υπέρ 28 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, ας το ελέγξουμε όμως. Πέρασε της ψηφοφορία. 28 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές. Πάλι νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Πέρασε της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. Φτάσαμε τώρα στο τέλος ε, στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 52 υπέρ, 5 κατά και 9 αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Κύριε Σιγητά. Είπα 52 υπέρ, 5 κατά, 9 αποχές. Δεν τα βλέπετε καλά. Jetzt haben wir noch eine schwierige, langwierige Abstimmung. Και τώρα έχουμε την έκθεση Παντσέρη. Δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Παντσέρη για να μην κάνει ακόμη μακροσκελέστερη αυτή τη διαδικασία. Υπέρ. Ή ε, πρέπει να το κάνουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 60 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στη συζήτηση της έκθεσης ε, για τα Ηνωμένα Έθνη. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Βαϊράινεν είναι ο εισηγητής. Το είχαμε αναβάλει από την προηγούμενη φορά. Θα του δώσουμε τώρα το λόγο. για να μας κάνει την παρουσίαση. Να πω ακόμη κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Αύριο, μεθαύριο μάλλον, στις 12, είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και στις 12 Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει και πάλι αυτή η έκθεση. 13 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και στην δεύτερη Ρωμέλεια του Νοεμβρίου θα ψηφιστεί. Συμφωνείτε με αυτό το χρονοδιάγραμμα? Συμφωνείτε και δίνω το λόγο στον κύριο Βαϊράινεν. Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκθεση νωρίτερα αλλά μετά δεν υπήρχε χρόνος για συζήτηση. Επομένως, θα επαναλάβω εντάχει την εισαγωγή μου. Η ιδέα μιας έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών προέκυψε το Σεπτέμβριο πέρσι όταν ο κύριος Κέβιν Βότκινς έκανε μία έκθεση ενός ευρωπαϊκού think tank ε, τα συλλογικά μας συμφέροντα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται παγκόσμιες λύσεις και τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται ευρωπαϊκή δράση. Ε, Τότε λοιπόν είχα προτείνει να γίνει μια ίδιας πρωτοβουλία για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Αργότερα το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης περιορίστηκε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών για το πώς μπορούμε καλύτερα να επιτύχουμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής μας. Ο περιορισμός αυτός δεν ήταν και τόσο σημαντικός ε, στην πράξη, διότι τα Ηνωμένα Έθνη μέσω του συστήματός τους ε, καλύπτουν όλες ε, τις πολυμερείς παγκόσμιες μορφές συνεργασίας. Αυτό το οποίο λείπει είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εκτός Ευρώπης και ομάδες χωρών εκτός Ευρώπης. Αλλά η έκθεση αυτή καλύπτει όλες τις ε, πολυμερείς ε, πτυχές παγκόσμιας συνεργασίας. Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε τρία στοιχεία. Πρώτα, παρουσιάζονται οι στόχοι εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των συνθήκων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ως βάση να εξετάσουμε τους στόχους και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τους στόχους αυτούς στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια υπάρχει μια εισαγωγή, σύντομη παρουσίαση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια ε, εν τέλει παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση περιλαμβάνει και κάποιες προτάσεις για την ενίσχυση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ε, να γίνουν κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επαναλαμβάνεται επίση η πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, δεν ε, θεωρώ προσωπικά ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ ρεαλιστική, αλλά επειδή πρόκειται για πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχω συμπαριλάβει και αυτήν στην έκθεση. Στη συνέχεια υπάρχει ιδέα σύστασης ενός νέου σημαντικού φορέα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ε, με τίτλο ε, Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θα καλύπτει όλες τις πολιτικές εκτός ε, των θεμάτων ασφαλείας, τα οποία ούτως ή άλλως χειρίζεται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η σύνθεση και το καθεστώς αυτού του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του Συμβουλίου Ασφαλείας, να έχει δηλαδή μόνιμα και τακτικά μόνιμα μέλη, τακτικά μέλη και εκπεριτροπής μέλη ε, προτείνω όμως να μην υπάρχει δικαίωμα ε, αρνησικυρίας στο Συμβούλιο αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης προτείνω να συσταθεί ένα μόνιμο κοινοβούλιο. Έχω ακούσει κάποιες επικρίσεις επ' αυτού. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα μπορούσαμε ίσως ε, να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό βάσει του οποίου θα έχουμε μια κοινοβουλευτική συνέλευση ως ένα πρώτο βήμα και μετά ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος να είναι η σύσταση ενός ε, ε, πραγματικού κοινοβουλίου. Είναι ιδεαλιστικός αυτός ο στόχος, αλλά πρέπει να είμαστε και ιδεαλιστές ε, όταν πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω οι πιο σημαντικές παράγραφοι στο κείμενο είναι οι παράγραφοι 12, 13 και 14, οι τελευταίες δηλαδή οι παράγραφοι, στις οποίες ε, χαιρετίζουμε την διοργάνωση σε συγκεκριμένες ομάδες, κλάστερς, ε, ε, των διαφόρων επιτροπών, δίνοντας στον αντιπρόοδο, είπα το εκπρέσωπο, την αρμοδιότητα της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τονίζεται ότι η παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου κλάστερ. Κατόπιν προτείνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με τον ίδιο συνολικό τρόπο και να οργανώσει τις εργασίες του αντιστοίχως. Ε, θεωρούμε ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να αναλάβει το συντονισμό όλων των τομέων πολιτικής ε, που άπτονται της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις αρμόδιες επιτροπές να γνωμοδοτούν σε κάθε θέμα και από εκεί και πέρα ζητάμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούν αυτή την προσέγγιση και να λογοδοτούν σε αιτήσια βάση για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορούμε κάθε χρόνο να διαμορφώνουμε άποψη για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση είναι διατυπωμένη κατά τρόπον ώστε να επικεντρώνεται στις ε, βασικές αρχές και στις βασικές γραμμές πολιτικής μας και ελπίζω οι τροπολογίες να μην υποσέλθουν σε πάρα πολλές λεπτομέρειες διότι υπάρχει μια ετήσια έκθεση για τα Ηνωμένα Έθνη ε, στην οποία τα ε, καθημερινά αν θέλετε θέματα ε, της πολιτικής με τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρονται. Επομένως εδώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε στις γενικές ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και να ενισχύσουμε και την παγκόσμια επιρροή μας εν γέννη. Αυτό ε, σε γενικές γραμμές ε, κύριε Πρόεδρε είναι το σκεπτικό του σχεδίου κειμένου και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας, να έχω και τις σχετικές τροπολογίες σας και από εκεί και πέρα να διαπραγματευτούμε για τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Συναντήθηκα με κάποιους από τους κοιόδης εισηγητές, έχω ζητήσει από όλους να παραστούν στη συνεδρίαση, αλλά δεν ήταν και τόσο επιτυχής η προσπάθεια. Θα έχουμε όμω χρόνο και στη συνέχεια να συναντηθούμε και να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, ε, αυτά από μένα. Προσβλέπω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριο Σπρέντα. Ο Αρνό Ντανζόν δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα. Παρουσιάζω λοιπόν την παρέμβασή του στη θέση του. Και εξάλλου συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις που θα ήθελε να διατυπώσει. Ο Αρνό θέλει καταρχήν να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεσή του και για το έργο του. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τον εισηγητή για να μπορέσει να βελτιώσει ορισμένες πτυχές της εκθέσεως αυτής. Γι' αυτό θα καταθέσει μια σειρά και από τροπολογίες με στόχο να ξαναεπικεντρώσει την έκθεση στα θέματα εξωτερικών υποθέσεων με το να τονίσει περισσότερο τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να μπορέσει να δώσει και μεγαλύτερη έμφαση στο να αντιμετωπιστεί αυτή η προβληματική από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θεωρεί ότι η έκθεση εστιάζει υπερβολικά στο στη δομή του ΟΗΕ και στην βιώσιμη ανάπτυξη και λιγότερο από ό,τι πρέπει στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξουν τροπολογίες επίσης, οι οποίες έχουν σε στόχο να αντιμετωπίσουν πιο ουσιαστικά τον κυρίαρχο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να έχει η Ένωση μέσα στα Ηνωμένα Έθνη και επίσης την υποστήριξη προς το προσωπικό του ΟΗΕ σε ενέργειες διατήρησης της ειρήνης. Θέλω να εκφράσω λοιπόν και την ικανοποίησή μου για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες θέσεις και επίσης για τις ε, αποστολές της Ομαλίας στο Μαλί και στο Μαλί Σαχέλ. Θέλω να εξάρω τον, τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ. Η έκθεση θα πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ στα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων και ιδίως στα πλαίσια της ε, διατήρησης της ειρήνης και σε αποσμένους εξειδικευμένους φόρεις. Πρέπει η έκθεση αυτή να παραμείνει πιστή στην επίσημη θέση του Κοινοβουλίου να έχει μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτό να αποτελέσει ένα στόχο μακροπρόθεσμο. Θέλει ο κύριος Ντανσόν να τονίσει ότι περιμένοντα μια τέτοια μεταρρύθμιση, τα κράτη-μέλη τα οποία παρακάθονται στο Συμβούλιο ασφαλεία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληροφορούν και τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι δραστηριότητε και τι θέσει του. και θα ήθελα επίση να υπογραμμίσει τη σημασία που επέχει το να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και κοινέ θέσει μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα κοινή εξωτερική πολιτική στα πλαίσια του ΟΗΕ. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να περνά από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η πρακτική κατά την οποία ο, η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι κάτι του Ηνωμένων Εθνών, είναι κάτι που υποστηρίζουμε. Αυτές λοιπόν οι απόψεις του Αρνοντανζόν και όπως σας είπα στην αρχή, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ένα ακόμα σημείο θα ήθελα να προσθέσω γιατί ξέρω ότι ο κύριος Βάιρινεν είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, στην οποία είμαι και εγώ μέλος, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ιδέα ενός Συμβουλίου για την βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να τροποποιήσουμε και την θεσμική ε, αρχιτεκτονική του φορέα αυτού για να τονίσουμε περισσότερο τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό να υπόκειται στο Συμβούλιο αυτό ο, η δραστηριότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΠΟΕ. Ευχαριστώ που με ακούσατε με τόση προσοχή. Ο πρόεδρος με χωρίς μικρόφωνο. Ε, Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πόστ, ε, ευχαριστώ την εισηγήτη καταρχήν. Η έκθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή βάση για τη συζήτηση και μπορεί να τονίσει τη σημασία που πρέπει ε, να έχει ο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μιλούν με μία και μόνη φωνή στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλου διεθνεί οργανισμού, ε, ιδίω για να τονίζουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνει στην μείση διάταξη το θέμα αυτό, ούτω ώστε συνεχώ να φροντίζουμε για την ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό θέμα στο διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ελπίζω ότι την έκθεση θα τονίζεται ο πιο ισχυρός ρόλος που πρέπει να παίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ε, Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε μια ξεκάθαρη εντολή όπου θα υπάρχει σαφώς και η συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω υποβάλει κάποια τροπολογία. όπου τονίζεται το ψήφισμα 1325 ε, που αναφέρεται στο ρόλο των γυναικών ε, σε καταστάσεις διενέξεων η διάσταση των φύλων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία της ε, μεταρρύθμισης και στο μέλλον θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ιδέα μιας γυναίκας στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων θα πρέπει επίσης να είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Σημειώνω ακόμη το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση του μορατόριου για τα χημικά όπλα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να μάχεται ε, για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και για τη μη διακριτική μεταχείριση. Χαιρετίζουμε επίση και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και στο πλαίσιο αυτή της έκθεση. Ε, το ότι έγινε η πρώτη ε, συνάντηση για τα δικαιώματα των ε, ΛΔΟΑΤ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το έγγραφο αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο παρέχει ε, έδαφος για συζήτηση για διάφορα θέματα, εκ των οποίων άλλα θα συζητήσουν περισσότερο και άλλα ε, λιγότερο στο μέλλον. Η έκθεση αυτή δεν μιλά για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγμή. Περισσότερο αποτελεί ένα σχέδιο προτινόμενων μεταρρυθμίσεων για τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι διαφορετικό θέμα και από τεχνικής πλευράς θα έλεγα ότι είναι πέραν τη εντολή που δόθηκε στον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Η ομάδα του ECR βεβαίω είναι υπέρ ε, του πολυμερούς επίπεδου, του πολύπλευρου επίπεδου στα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως ε, κάθε χώρα δεν μπορεί να ε, προχωρεί μόνη της και γι' αυτό υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και για την ε, πρόληψη κρίσεων και για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την παγκόσμια υγεία κλπ. κλπ. Αλλά αυτή η έκθεση δεν θα έπρεπε να τονίζει αυτά τα θέματα τα οποία πραγματεύεται τώρα. Η ομάδα μας γνωρίζει ότι βεβαίως και χρειάζονται κάποιες μεταρρυθμίσεις που κάποια στιγμή θα προκύψουν, αλλά δεν ε, ε, ε, συμφωνούμε με το να εγκαταλείψουμε τη θέση των δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και στο πλαίσιο των συζητήσεων 5 συν 1. Ε, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η Γερμανία πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο ως μόνιμο μέλος ε, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας μαζί με την Ινδία και την Ιαπωνία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει σχετικά επιχειρήματα. Εδώ συζητήσαμε και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού, το Συμβούλιο του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι ε, ένα νέο θέμα και συγχαίρω τον εισηγητή για την ε, νέα αυτή πρόταση. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος για τη σκοπιμότητα. Με βάση τους τρεις πυλώνες, ε, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό, έχουμε στα Ηνωμένα Έθνη κάποιους τομείς που μπορούν να ενδυναμωθούν αντί να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, ένα νέο συμβούλιο με νέες εξουσίες και αρμοδιότητες. Δεν νομίζω ότι η ομάδα του ΙΣΙΑ θα δεχτεί αυτή την πρόταση ως έχει. Πάντω συγχαρητήρια στον εισηγητή για την προσπάθεια προώθησης ε, καινοτόμων ιδεών. Προς το παρόν όμως η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών γενικότερα ε, βρίσκεται σχεδόν σε στάδιο παράλυσης ε, γιατί κάθε φορά που θα προταθεί ένα νέο μέλος μια άλλη χώρα στην ίδια περιφέρεια θα βρεθεί να έχει αντιρρήσεις κάτι το αναμενόμενο εξάλλου στο τωρινό πλαίσιο. Ενδιαφέρουσα η έκθεση λοιπόν αλλά η ομάδα μου φοβάμαι ότι δεν θα υποστηρίξει κάποια τμήματα της έκθεσης που προτείνονται. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω την έκθεση αυτή που περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέρουσες ιδέες. Θέλω όμως να σας προειδοποιήσω να μην μετατρέψετε αυτή την έκθεση σε κάτι το οποίο προτείνει μια ριζοσπαστική αλλαγή του συστήματος του ΟΗΕ. Κάποιες από τις ιδέες που αναφέρατε θα ήταν χρήσιμο να συζητηθούν περισσότερο στην ομάδα εργασία τη ΑΦΕΤ και τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ. Αυτή η ομάδα εργασία έχει δύο χρόνια να συνεδριάσει. Νομίζω όμω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε κάτι τόσο μεγαλόπνο. Στην έκθεση αυτή χαιρετίζω την ε, αναφορά στο ΟΗΕ ως υπερασπιστή της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω διάφορε προτάσει, τις, θα τις απαριθμίσω, απλώς θέλω να αναφέρω κάποιες ιδέες. Νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει γενικά την διεθνή δικαιοσύνη μέσω του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Περιφερειακών Φορέων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει επιτυχεί η Ευρώπη για την ε, <clears throat> τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα για άλλες περιοχές που συμμετέχουν στα Ηνωμένα Έθνη. Αναφέρω επίσης ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται και στην ειδική έκθεση του Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΗΕ σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να τονίσει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια πιο αποτελεσματική και ε, προσιλωμένη δράση για την υποστήριξη των ενεργειών του ΟΗΕ η ύπατη εκπρόσωπος και οι αρμόδιες αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές αστάθειας θα πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ορατότητα και αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρετε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κέριος εταίρος των Ηνωμένων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Νομίζω το είπε και η κυρία Μογγερίνη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την πρώτη της ε, την πρώτη δήλωση σε σχέση με την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΗΕ, ενθαρρύνοντας μας να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτή <clears throat> εταιρική σχέση. Τόνισε επίση η έκθεση το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα, τον έλεγχο εξοπλισμό και η κυρία Φώση έχει κάνει κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να χαιρετήσουμε την έγκριση συμφωνίας Άμστρατ από το Συμβούλιο Ασφαλείας και επίσης η, μάλλον η συνδική για, για το εμπόριο όπλων από την Γενική Συνέλευση και επίσης να προωθήσουμε τις σχετικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω περιοριστεί μονάχα σε μερικές από τις τροπολογίες που θα καταθέσω. Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω έχει να κάνει με την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου θα ήταν καλό να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υπάρχουσες αυστηρές ερμηνείες του διεθνούς δικαίου που λένε ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και ιδίω το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τα υπόλοιπα μπορώ να σας τα δώσω γραπτά. Ευχαριστώ λοιπόν, χωρίς μικρόφωνο πάλι, δίνει το λόγο στον επόμενο μιλητή. Ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα αυτή η έκθεση και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά και όσον αφορά τη δική μας τη θέση στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και ε, τις αδυναμίες ε, της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το οποίο μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η πρόταση ε, η οποία κυκλοφορεί άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό όσον αφορά τη δυνατότητα ε, τα Ηνωμένα Έθνη ε, να μας παρηχωρήσουν μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να παραμένει εκρεμές αυτό το ζήτημα για το τι ακριβώς ε, θα γίνει στο μέλλον ε, για τις ε, θέσεις που καλύπτουν αυτή τη στιγμή η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας, τον οποίο θα αποτελείται αντί από κράτη, από περιφερειακές οργανώσεις όπως είμαστε εμείς, η Αφρικανική Ένωση ή η ΑΣΕΑΝ. Επίσης, θα ήταν ίσως χρήσιμο να εξετάσουμε και την πιθανή μεταρρύθμιση αυτού που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας, ε, αν βέβαια υπάρξει και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το δικαίωμα δηλαδή του βέτο. Ε, ξέρουμε ότι ορισμένες φορές όταν δεν υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις, πολύ δύσκολα μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μια πρόταση από πλευρά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει η δυνατότητα μιας ειδικής πλειοψηφίας. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της ύπατης εκπροσώπου και το την οργάνωση σε κλάστερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη νέα θητεία είναι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρονται. Πρόκειται για ένα θετικό στοιχείο το οποίο στο μέλλον ίσως θα μας επιτρέπουν να έχουμε και ένα καλύτερο συντονισμό αλλά θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και κάτι περισσότερο από έναν απλό συντονισμό, να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή κυρίως στην εμπορική πολιτική σε σχέση με τις υπόλοιπε εξωτερικές πολιτικές. Ένας πιο ισχυρός εκπρόσωπος ίσως θα είναι ένα καλό τρόπος να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε η εμπορική πολιτική η οποία θα είναι ε, στην υπηρεσία της γενικότερης εξωτερικής πολιτικής και όχι το αντίστροφο θα βασίζεται και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και ίσως και μια ευφυούς και σόφρονος ε, χρήσης της ε, soft power. Αυτά είναι μια σειρά αποσκέψεις ε, που αναφέρονται σε ένα μέλλον που ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθούν, αφορούν τη μεταρρύθμιση της Γενικής Συνέλευσης, ε, το να γίνει ένα ε, πιθανό παγκόσμιο κοινοβούλιο, αλλά έτσι ίσως θα μπορούμε να έχουμε άμεση έκφραση της βούλησης των διαφόρων λαών. Ξέρουμε βέβαια ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί πάρα πολύ δύσκολα, για να μπορεί να είναι αξιόπιστο ένα τέτοιο κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να εγγυάται και την διεξαγωγή ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών σε όλα τα κράτη που θα συμμετέχουν, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μάλλον ουτοπικό και ε, στην καλύτερη των περιπτώσεων σε πολλές χώρες ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές παρατυπίες και προβλήματα για διεξαγωγή αμερόληπτων εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσω τροπολογιών μας θα φροντίσουμε να κάνουμε κατάλληλες παρατηρήσεις που θα είναι αντίστοιχα των όσων μόλις εξέφρασε. Ευχαριστώ πολύ. Μακάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα μιλήσω μονάχα εν συντομία. Να αναφέρω ότι στη Συνταγματική Επιτροπή η εισηγήτρια για μια γνωμοδότηση σε σχέση με την έκθεση αυτή έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες στην αντίστοιχη δική μου έκθεση. Είναι πλήρης η έκθεση του Φιλανδού συναδέλφου, αλλά υπάρχει ένα σημείο για το οποίο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι οι κυριότεροι χρηματοδότες του ΟΗΕ και αναφερόμαστε επίσης και στην, στα πλαίσια της, της ε, πρωτοβουλίας Delivering as One να βελτιώσουμε την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παρέχει όλα αυτά τα μέσα στα Ηνωμένα Έθνη και ζητούμε και από το ΟΗΕ όπως και από την Κομισιόν να αναφέρεται και να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ηνωμένα Έθνη. Sorry. Ah, thank you. Uh, I, would like to thank Και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας για την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω σε γραπτή μορφή αυτά τα οποία λέμε εδώ, ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν είναι μοναχα ένα κέριο θέμα, όχι μοναχα για τη λειτουργία του ΟΗΕ, αλλά για την αποτελεσματικότητα του ΟΕ και κυρίως για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να έχει μια έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Μόνο έτσι μπορούμε να συντονίσουμε με οργανωμένο τρόπο τις ενεργείες μας. Δεν είναι για ένα ή δύο κράτη-μέλη, είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την ε, κρίση που αφορά τη Συρία, γιατί δεν έχει λειτουργήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και φυσικά πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η δυνατότητα ανησυχηρίας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πιο περιοριστική, δεν θα πρέπει μόνο μια χώρα με ένα βέτο να μπορεί να εμποδίσει τη δράση του πρέπει να είναι δύο ή τρει. Και νομίζω ότι προφανώς είναι α, αναντικατάστατη η λειτουργία του ΟΗΕ, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και το ρόλο της τη Αρμοστία για τους πρόσφυγες. Όπως είπε ο κύριος Κουτέρε το πρωί, Εμεί δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το διεθνέ δίκαιο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την προ όθηση και την επικράτηση του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να παραβιάσουμε στο δίκαιο και σε σχέση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα από τα κάτι μελη μας η Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιεί τα μη επανδρομένα αεροπλάνα για στοχευμένους φόνους. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώπιον αυτού του θέματος Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σταθούμε στο θέμα αυτό. η είπατε εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη θα πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη προ την κατεύθυνση αυτή. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτέλου εκδίδει μια έκθεση για τα θέματα αυτά. Πρέπει να ζητήσουμε όμω από την κυρία Μογκερίνη να έρθει αντιμέτωπη με τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε πόσο δύσκολη η κατάσταση για την ε, εμπιστοσύνη τη κοινή γνώμη έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο μέσα από περισσότερη ένωση μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει τα κράτη-μέλη να επομιστούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εμείς μπορούμε να την πετύχουμε αν συμφωνούσαμε για το πώς θα μοιραστούμε μεταξύ μας την εκπροσώπηση στον ΟΗΕ και έτσι να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. κύριο Κάρβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συγητή. Έχουμε και το μελλοντικό δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει ιδέε για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών. Θέλει να αναλάβει περισσότερα ενία και περισσότερη εξουσία, προσπαθεί να αυξήσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος των κρατών μελών και προτείνει μάλιστα και μια παγκόσμια κυβέρνηση που δείχνει ότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστής. Και επίσης ε, θέλει να ξοδέψει πολύ περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων για πιο ακριβές ε, ε, τελετές χωρίς λόγο. Και προτείνω λοιπόν, ε, όταν προτείνει να τελειώνουν ε, με τις θέσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο, μόνιμο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να έχουμε μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα για να έχουν αυτές τις θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και είναι πηγές ε, ειρήνης και σταθερότητας από τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, όπω γνωρίζετε, συχνά διαφωνούν, αλλά έχουν πολύ μεγάλη πείρα στο Συμβούλιο Συμβούλιο Ασφαλεία και αυτό αντανακλέκεται εθνικά του συμφέροντα, κάτι το οποίο δεν υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίση συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γίνεται σεβαστό στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Πώ μπορεί να είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να στερηθεί δύο έδρε αντί για μία, για να ε, ε, διασφαλίσει περισσότερη διεθνή ασφάλεια στα κράτη-μέλη. Δεν τα υποστηρίζουμε και δεν νομίζω ότι θα τα υποστηρίζει και η εκλογική μου περιφέρεια. Όσον αφορά τι ε, ε, συμμετοχές ε, στα Συμβούλια ασφαλεια Ασφαλεία, αυτοί συμμετείχαν πολλά κράτη-μέλη. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλεία λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά από τότε που ξεκίνησε και ε, παρά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παγκόσμιο παίκτη σε θέματα ασφαλείας και δεν νομίζω ότι μπορεί να προσδώσει περισσότερη ασφάλεια Υπάρχουν διάφορες ε, διαμάχες, όπως για παράδειγμα τα όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια, που είναι παράδειγμα που μας αποδεικνύουν ότι πραγματικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί να πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοια θέματα, σε παγκόσμιες κρίσεις. Όσον αφορά τις προτάσεις για τον προπολογισμό, είναι άλλο ένα παράδειγμα για το, την απώλεια κυριαρχία των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλαμβάνει ευθύνε οι οποίε είναι περιττές. Δεν θα έπρεπε να αναλαμβάνει τέτοιε ευθύνε. Υπάρχει μια σαφή διαδικασία για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν πρεσβεία σε μια χώρα. Δεν χρειάζεται ε, ε, ένα γραφείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι μια άλλη περίπτωση περί των δαπανών, περί της ε, ανάμειξης σε ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο ρόλο και να δικαιολογήσει την ύπαρξή της. Και ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και νέες οργανώσεις όταν δεν χρειαζόμαστε καμία οργάνωση. Στο σημείο 8 προσπαθούμε να έχουμε κάποιες επιτυχείς οργανώσεις όπως για παράδειγμα την Παγκόσμια Τράπεζα υπό τη σκέπη μας. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δεν έχει μάθει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της. Το σημείο 9 τονίζει ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ηρωνικό το να προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε εμείς τα πράγματα. Νομίζω ότι είπα αρκετά κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κόβατσεφ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για το ενδιαφέρον αυτό σχέδιο έκθεσης. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πρέπει να τονίσουμε τον ε, έντονο ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα θέματα ψηφισμάτων, ιδίως τώρα με τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα κάνουν κάτι και αυτό έχει μειώσει πάρα πολύ την ε, εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Δεύτερον, να προωθούμε μια μεταρρύθμιση των ΗΕ Εθνών ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εμεί και το Συμβούλιο για τι μεταρρυθμίσει που επιθυμούμε. Στο σημείο 14 του ψηφίσματο που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο, ζητάμε από το Συμβούλιο να υποβάλει ετησίω έκθεση στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε και ε, για τον κατάλογο μεταρρυθμίσεων. Τι θέλει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις μεταρρυθμίσεις ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρουμε ότι είναι απειρχιωμένος ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από τόσα χρόνια που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945 αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει η βούληση να δεχθούν νέα μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή να αλλάξουν οι κανονισμοί όσον αφορά το δικαίωμα άρνηση κυρίας. Άλλο ένα σημείο θέλω να αναφέρω για την εκλογή ε, του επομένου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας ότι έχει φτάσει η στιγμή κάποιος από την Ευρώπη να αναλάβει και γιατί όχι μια γυναίκα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλανμόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια φιλόδοξη έκθεση, περιλαμβάνει μια σειρά από νέες προτάσεις και θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη διότι δεν αναφέρεται μόνο στην ανάγκη να βελτιώσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά επίσης και προτείνει κάποιες μεταρρυθμίσεις για τα Ηνωμένα Έθνη. Και νομίζω ότι επικεντρώνεται πολύ σε αυτή τη δεύτερη πτυχή, η οποία μάλλον είναι πιο ευρεία από τον τίτλο της έκθεσης και εδώ θα ήθελα να είμαι λίγο επικριτικές. Αυτό το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο είναι μια ιδέα κατά την άποψή μου την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι, μεν είναι κάτι το οποίο είναι μακρόπνο, όπως λέει και η έκθεση, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τέτοιες ιδέες και δεν νομίζω αν, ότι είναι η κατάλληλη θέση, η, η πιο κύρια θέση της έκθεσης, το να δημιουργήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο. Τον αναφέρεται ως πρώτο σημείο ε, υποδεικνύει ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, ε, ιδέες. Δεν πιστεύω βέβαια ότι ισχύει κάτι τέτοιο γιατί μετά λέγεται ότι είναι μακρόπνο όραμα. Συμφωνώ με την ιδέα της μόνιμης θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι μακροπρόθεσμα. Ε, και νομίζω ότι αυτό ε, καλύπτει και την πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, μπορεί να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Μια άλλη πτυχή τώρα Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλά ε, αν ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 2013 έγινε μια πολύ σημαντική ε, μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν ο ΙΕ θέλει να δημιουργήσει ένα νέο τόσο φιλόδαξο όργανο. Ε, και για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω με ποια λογική θα πρέπει να έχουμε ένα συμβούλιο, δηλαδή τον αναχρονισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας, να τον επαναλάβουμε σε ένα άλλο συμβούλιο με μόνιμα μέλη. Ε, αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, συστήθηκε το 1945 και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα γιατί σήμερον ημέρα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πέραν αυτού υπάρχουν και προβλήματα διακυβέρνησης για όσους εργάζονται στον ΟΗΕ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το Συμβούλιο γενικά είναι καλή ιδέα. Και τέλος, και με αυτό ολοκληρώνω, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το λέει και ο εισηγητής στο τέλος, αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω ακόμα περισσότερο σε αυτό, ότι το Ηνωμένα Έθνη είναι ένα από τα αποτελεσματικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτυχάνει τους στόχους τους. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συντονίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Και εγώ νομίζω ότι ε, ε, ε, έτσι θα έπρεπε να γραφτεί. Υπάρχει και το άρθρο 34 που το προβλέπει αυτό. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπεται τα μόνιμα μέλη να υπερασπίζουν τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφερόμαστε και στο ρόλο συντονισμού, της υπάτης εκπροσώπου και το Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια συντονισμένη δράση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με μια φωνή και τα κράτη-μέλη να δρουν συντονισμένα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση που έχει πολλέ ε, πολλές ιδέες, κάποιες από αυτέ καινούργιε. Ευχαριστώ και πολύ. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο, συνηθίζει. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Λέω και ο Γκάλερ, σε ένα σημείο μονάχα θα εστιάσω. για την πιθανή μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν θέλω να κάνω οικοτολογίες, αλλά όταν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματιστικά και να θεωρήσουμε δεδομένο ότι μια τροποποίηση του καθεστώτους των πέντε μονίμων μελών που έχουν και το δικαίωμα του βέτο δεν φαίνεται να είναι κάτι το εφικτό. Δεν έχουν βέβαια το ίδιο την ίδια δύναμη που είχαν το 1945 και τα πράγματα αυτά δεν θα μπορούν να παραμένουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι απαραίτητο χώρες όπως η Ινδία να έχουν και αυτές μια μόνιμη έδρα στο Συμβουλίο Ασφαλείας και βρίσκω την ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα να μπορούν οι περιφερειακοί οργανισμοί να έχουν μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να έχουν βέτο ή όχι. Αν πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόσθετη ε, έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Αφρική ή η ΑΣΕΑΝ, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τότε να μπορεί να ψηφίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας μόνο αν υπάρχει ομόφωνη συμφωνία. Και έτσι θέματα εξωτερικής πολιτικής μπορούν να προαποφασίζονται ώστε να μπορεί να ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και τα δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν πια τη δυνατότητα να ψηφίζουν χωριστά και μεμονωμένα. Απλώς θα έχουμε τριπλασιάσει λοιπόν έτσι το ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε τον επικοδομητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά θετικά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και έτσι λοιπόν θα ήταν μια πολύ ελκυστική μέθοδος να ψηφίζουμε όταν έχουμε ακριβώς την ε, ε, ομοφωνία. Και τότε οργανώσεις περιφερειακές ε, από την Λατινική Αμερική ή από την Ασία, από την Αφρική μπορούν και αυτές να συμμετέχουν υπό τον όρο να είναι ομόφωνες. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εδώ Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες ιδέες που έχουν παρουσιάσει, τα ενάφησματα που έχουν παρουσιάσει στις παρεμβάσεις τους. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας και τις συζητήσεις με τους κοιόδης συζητητές των διαφόρων ομάδων. Απλώς θέλω να πω κάτι σε σχέση με τη βασική ιδέα που διατρέχει την εκθέσή μου. Προφανώς ο στόχος είναι να ενισχύσουμε το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Χάρη στον καλύτερο συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο όλων των εμπλεκομένων και όλων των πολιτικών μέσα στο σύστημα του ΟΗΕ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και το Συμβούλιο Αηφόρο Ανάπτυξης. Δεν είναι μια νέα ιδέα, και εγώ ήμουνα στο Ρίο στην ε, συνδιάσκεψη του 1992 όταν τέθηκε για πρώτη φορά. Στα Ηνωμένα Έθνη οδήγησε σε μια ισχνή συμβιβαστική λύση και τίποτα το ουσιαστικό. Η ιδέα λοιπόν του να έχουμε αυτό το νέο συμβούλιο είναι πολύ σημαντική και εξάλλου θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με τρόπο αποτελεσματικό να επηρεάσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι δύσκολο να έχουμε μια πιο ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση γιατί η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν να παραδώσουν τις έδρες τους, ούτε και άλλες μεγάλες δυνάμεις φυσικά είναι έτοιμες να δώσουν μια πρόσθετη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό χωρίς ε, δυνατότητες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Εγώ λέω φυσικά στην έκθεσή μου ότι πρέπει να έχουμε μια έδρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό στο ορατό μέλλον. Αν έχουμε όμως το Συμβούλιο Αϊφόρου Αναπτύξεως, χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία που θεωρώ ότι πρέπει να έχουν και μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας μπορούν να είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και μέσω αυτού του Συμβουλίου να αυξήσουν την επιρροή τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα είναι ένα από τους κέριους παίκτες σε αυτό το νέο Συμβούλιο. Αυτή η αρχιτεκτονική λοιπόν που προτείνω εξυπηρετεί τους στόχους αυτής της έκθεσης για το πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής μέσω του συστήματος του ΟΗΕ και μέσα από ένα καλύτερο συντονισμό των πολιτικών μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω λοιπόν όπως σας είπα στις τροπολογίες των συναδέλφων που και τελικά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Πολλά θα μπορούσα να σχολιάσω. Ίσως όμως είναι καλύτερα να σταματήσω εδώ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε άλλο ένα σημείο για να ενισχύσουμε την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει σε πολλούς τομείς στα προγράμματα των ΗΠΑ σε μεγάλο βαθμό και πρέπει να βελτιώσουμε την ορατότητά τη, αλλά γιατί κανείς δεν γνωρίζει τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε εμεί οι ίδιοι δεν το γνωρίζουμε, εκτό από του ίδιου οι οποίοι συμμετέχουν σε, αυτέ τι δραστηριότητε. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν ε, ε, τον τρόπο, να, δώσουμε, ε, να βρούμε το μέσο, να δώσουμε μια όθηση στην ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακόμη και για τους πρόσφυγες ε, βλέπουμε ότι υπάρχει το όνομα των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, υπάρχει το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτών, αλλά δεν υπάρχει ακόμη και το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διεξάγουμε δράσεις ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας το έχουμε κατά νου αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ας σταματήσουμε για λίγα λεπτά ή έχουμε κάτι άλλο να μην διακόψουμε. για την κατάθεση τροπολογιών ε, μεθαύριο 12 το μεσημέρι, 17 Σεπτεμβρίου. 15 λεπτά διάλειμμα να περιμένουμε τη Helga Schmidt. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη συμφωνία με το Ιράν.